των δύο φύλων. Σχόλιο από αυτού. Ο ορισμός λοιπόν εγκρίνεται. Επίσης από τις αρμόδιες ουγγρικές αρχές ε, μου έχει φτάσει έτοιμα για την άρση ασυλίας του κυρίου Ταμάς Ντόιτς. Βάσει του αρθρού 6 παράγραφος 3 το αίτημα αυτό θα βάσει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που είναι και η αρμόδια επιτροπή για το θέμα. Η κυρία Μαγδαλένα Άλβαρες τώρα μου ανακοίνωσε γραπτά ότι ορίστηκε αντιπρόεδρος